και στις ε, ε, δυσμεύσεις των επιχειρήσεων. Αν θέλουμε να γίνουν πραγματικά βήματα προς το μέλλον, δεν θα πρέπει να σκεφτούμε μόνο τις δημόσιες αρχές, αλλά να σκεφτούμε και όλες τις υπόλοιπε πτυχές. Ευχαριστούμε κύριε Ντελάγκε. Ολοκληρώνουμε λοιπόν αυτό το σημείο. Να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές. Στη συνέχεια έχουμε τις παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού. Καταρχάς, ο κύριος Ιτουργκάιφ Αγγούλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας διαβιβάσω ένα μήνυμα από τον Ιζουάλντο Παγιά, ο οποίος έχει λάβει ε, βραβείο Σαχάρο. Αγαπητοί φίλοι, ο λαό τη Κούβα χρειάζεται αλλαγέ. Θέλει να δώσει ένα νέο, μια νέα όθηση στη ζωή του ή να ξεχάσει το μίσο, ε, την ε, καταπίεση και το φόβο θα πρέπει να ανοίξει η οδός της προόδου προς όλες τις κατευθύνσεις. Θα πρέπει να γίνουν αλλαγές οι οποίες ε, αλλαγές δεν επιβάλλονται μέσω νομοθεσίας, αλλά αυτή τη στιγμή ο Πρόεδρος διακόπτη δεν ακούει τη διερμηνία στα αγγλικά. Θα μπορούσαμε, κύριε Τουργκάης, θα ήθελα να μηδενίσετε και το χρόνο, λέει ο κύριος Τουργκάης. Και λίγο πιο αργά να μιλάτε, ζητά ο Πρόεδρος. Θα ήθελα να σας διαβάσω ένα μήνυμα λοιπόν από τον κύριο Παλιά, ο οποίος έχει λάβει βραβείο Ζαχάροφ από το Κοινοβούλιο. Ο λαό τη Κούβα χρειάζεται αλλαγέ. Χρειάζεται να μπει σε ένα νέο στάδιο τη ζωή του και να ξεχάσει το μίσο, τη βία, την καταπίεση, τα ψέματα και το φόβο. Θέλει να ξεκινήσει το δρόμο της προόδου προς όλες τις κατευθύνσεις και να γίνουν και οι σχετικές αλλαγές. Οι αλλαγές, ναι μεν δεν επιβάλλονται μέσω νομοθεσίας, αλλά ήδη ε, βρίσκονται στην καρδιά των κουβανών. Θα πρέπει να γίνουν σεβαστά τα πολιτικά τους και δικαιώματα, θα πρέπει να υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες, ε, ελευθερία του συναθρίζεσαι και του... Ε, συνεταιρίζεστε και θα πρέπει να μπορούν να ταξιδέψουν και σε άλλε χώρε. Θα πρέπει να αλλάξουν τα δικαιώματα, διότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν δικαιώματα οι Κουβανοί. Πολλέ φορέ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καταδιώκονται γιατί προσπα... προασπίζονται τα δικαιώματα των Κουβανών και βρίσκονται κλεισμένοι στι φυλακέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα Ένωση συγγνώμη, θα πρέπει να βοηθήσει αυτή τη θέση και θα πρέπει να παραμείνει ε, στη βοήθεια των Κουβανών. Υπάρχουν πάρα πολλές πρωτοβουλίες ε, και ε, ο λαός της Κούβας προσπαθεί να επιτύχει αυτές τις αλλαγές. Υπάρχουν πρωτοβουλίες τις οποίες θα πρέπει να υποστηρίξουμε κι εμείς γνωρίζοντας ότι υπάρχει μια κοινή θέση διότι θα πρέπει να υπάρχει και κοινή αντιμετώπιση του θέματος. Ευχαριστώ. Η κυρία Φλασίκοβα Μπένεβα για ένα λεπτό. ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι εξίσου σημαντικός όπως η καταπολέμηση της βίας. Συνεπώς, εάν ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει αστεία για τον Χίτλερ δημόσια μέσα ε, σε ένα πλαίσιο ε, θετικό, αυτό ο λόγος πρέπει να διαψευστεί, πρέπει να αντικρουστεί, διότι ε, δεν είναι ένα ηγέτης μιας δημοκρατικής ελεύθερης κοινωνίας και θα ήθελα να πω στον κύριο Μπερλουσκόνη ότι τα ε, γελία αστεία του δείχνουν είτε ότι έχει τρελαθεί είτε ότι δεν σέβεται τους δημοκράτες. Η κυρία Αλφάνο για ένα λεπτό παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, η Ιταλική εφημερίδα Ελφάτο Κοτουντιάνα δημοσίευσε το Σάββατο ένα κείμενο του πρώην μαφιόζου από το Παλέρμο, του Τσιβίνο, ο οποίος έλεγε ότι ο Μαρτσόλο ε, και ο ε, και ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη ήταν ε, παιδιά της ίδιας ομάδας, ανήκαν δηλαδή και οι ίδιοι στη μαφία. Αυτό το έγγραφο φτάνει στην εισαγγελία όταν μαθαίνουμε και την αλήθεια για τις ε, ε σφαγές που έγιναν το 1992, στην οποία πέθαναν δύο δικαστές, μεταξύ των οποίων και ο κ. Μπορσαλίνο όπως φαίνεται, από εκεί δημιουργήθηκε και το κόμμα του Πρωθυπουργού, του Φόρτσα Ιτάλια, ε, από έναν άνθρωπο ο οποίος καταδικάθηκε σε 7 χρόνια για τη μαφία και είναι ακόμα γερουσιαστής ε, στην Ιταλία. Ο Άντζελο Βασάλο, ο οποίος δολοφονήθηκε από, το, από την Καμόρα ε, και η ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο προσπάθησε να καταπολεμήσει τη μαφία και ζητήθηκε και από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών να γίνει κάτι για το, να συζητηθεί το θέμα τη Μαφία. Πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι πλέον τοπικό, είναι παγκοσμιοποιημένο και αφορά αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση ενό κράτου μέλους. Ο κύριο Τρεμόπουλο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζετε ότι, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι οι χώροι πρασίνου έχουν ζωτική σημασία για το αστικό περιβάλλον μάλιστα οι ειδικοί απαιτούν 7 έως δέκα τετραγωνικά μέτρα ανακάτοικο όσο δηλαδή και ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. οι, οι μεγάλες ελληνικές πόλεις όμως ασφικτιούν σήμερα με μόλις το 25 έως το 35% αυτών των απαιτήσεων και χρειάζονται επιγόντω πολλαπλάσιους χώρους πρασίνου. Μια προφανής λύση είναι να διατεθούν για πράσινο τουλάχιστον οι υπάρχουσες δημόσιες εκτάσεις Τέτοιε είναι το πλήθο των στρατοπέδων που υπάρχουν έχουν εγκλωβιστεί μέσα στι ε, πόλει, αλλά και το πρώην αεροδρόμιο τη Αθήνα στο ελληνικό. το μνημόνιο τη ελληνική κυβέρνηση με την κομισιόν και το Διεθνέ νομισματικό ταμείο στη σελίδα 28 προβλέπει την επανεξέταση τη αξιοποίηση δημόσια περιουσία με στόχο την αποπληρωμή του δημόσιου χρέου. αν οι περιορισμένε εφεδρείε δημόσια γη διατεθούν τελικά για το σκοπό αυτό το περιβαλλοντικό ισοζύγιο των ελληνικών πόλεων θα επιβαρυνθεί δραματικά και θα υποθηκεύσει το μέλλον. όλες οι ευρωπαϊκές πολιτικές για το αστικό περιβάλλον αναιρούνται από πέντε μόνο λέξεις ενός εγγράφου που επιβάλλεται σε χώρα μέλος από την ίδια την επιτροπή. ρωτώ μπορούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να δεχθούν κάτι τέτοιο; Ναι, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η κοινή γνώμη της Πολωνίας λυπάται για την έρευνα που γίνεται σχετικά ε, με, το, με την, ε, το ατύχημα ε, το αεροπορικό διότι λυπάται πάρα πολύ διότι η ρωσική πλευρά δεν διαβιβάζει τα έγγραφα τα οποία χρειάζονται και καθυστερεί όλη η έρευνα του θέματος. Θα έπρεπε η έρευνα αυτή να γίνει διεθνή ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσουν να επηρεάσουν την όλη έρευνα να επισπευστεί θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση πάνω στην ρωσική πλευρά, διότι χωρίς διεθνή πίεση και πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα υπάρξει καλή έρευνα σε σχέση με το όλο αυτό θέμα. Ευχαριστώ. Κύριος Περέρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, υπάρχει η κερδοσκοπία και μετά από τα μέτρα τα οποία επιβλήθηκαν στις χρηματαγορές ε, τώρα ε, έχουμε την επιβεβαίωση ότι όλα θα συνεχιστούν ότι τα πράγματα θα μείνουν ως έχουν η τα χρηματοοικονομικά παράγωγα οι αγορές προθεσμίες θα συνεχίσουν συνεχίσουμε με τις ίδιες μεθόδους, δεν θα αλλάξει ε, το θέμα της φορολογίας και όλα αυτά θα επειδή παρόλες ε, τις ε, ε, επιβολές λιτότητος εις τους εργαζόμενους που τους επευλήθη όλη την Ευρώπη και είναι προφανές στη Πορτογαλία, στη Γαλλία, στην Ελλάδα όλοι οι εργαζόμενοι ανθίστανται στη μέτρα που επιβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Μπάχμαν είναι ο πρώτος ο οποίος ε, έρχεται με τα χρώματα του κόμματός τους. Ε, χαρά δικιά μου κύριε Πρόεδρε. Φαίνεται ότι ο Νίκ Λέγ, ότι αντιπρόεδρος ε, της κυβερνήσεως στην Αγγλία θα ζητήσει να εφαρμοστεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και να μπορέσουν να ψηφίζουν και οι φυλακισμένοι ε, και ελέγχθη ότι θα ήταν ε, ε, ατυχές εάν υπήρχε πλήρης άρση και δεν εξήγησε ε, γιατί παραδείγματος χάρη είναι καλύτερο να μπορεί να ψηφίσει ένας κλέφτης αντί για ένας δολοφόνος. Θα μπορούν δηλαδή τα άτομα αυτά να εκλέγουν και τους νομοθέτες και πρέπει να σας πω ότι στο δικό μας κόμμα θα δεσμευτούμε ότι θα άρουμε μία τέτοια ε, μία τέτοια ε, νομοθετική ρύθμιση αναλόγως ποιος είναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Μόλτσερ. Ε, θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει περιοχή Φεριούλη, Βενετίας και Κροατίας όπου υπάρχουν ε, ιστορικές αντιφάσεις όπου προσπαθούμε να μπορέσει να υπηρετήσουμε επιβιώσει η γερμανικής προελεύσεως μειοψηφία του πληθυσμού στην Σλοβενία αλλά όταν χρειάστηκε να υπάρξει ε, μία ψηφοφορία ε, το αποτέλεσμα ήταν υπέρ της Αυστρίας ε, σε παλαιότερη ε, περίοδο και αυτή τη στιγμή υπάρχει μία κατάσταση η οποία δεν είναι θετική και προσπαθούν να επαναφέρουν την παλαιά Γιουγκοσλαβία. Ευχαριστώ κύριος Νικολέσκου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επισημάνω ένα πρόβλημα πάρα πολύ σημαντικό στην Ρουμανία, το οποίο όμως έχει προσλάβει διάφορες μορφές σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια σοβαρή κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο τις μικρόες και μισές επιχειρήσεις, κυρίως στο πλαίσιο της κρίσης. Το Εθνικό Συμβούλιο για τις Μικρομεσές κρίνει ότι οκτώ έως 10 επιχειρήσεις της 100 που έλαβαν χρηματοδότηση ευρωπαϊκή ε, αρετούνται των σχεδίων τους διότι δεν μπορούν να καλύψουν το υπόλοι, την υπόλοιπη χρηματοδότηση. Είναι κρίμα. Θα πρέπει όλοι ε, να προσδιορίσουμε νέα μέτρα υποστήριξης για τις μικρομεσαίες επειδή 70% του εργατικού δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης απασχολείται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Τίκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε λίγο θα αρχίσει η εξιαλόγηση της πορείας 2007-2013 του πολιετούς πλαισίου για μια συνεργασία διοργανική για να υπάρξουν λύσεις για την άμβλυνση των συνεπειών της κρίσης. Ταυτόχρονα η θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας και η στρατηγική 2020 προσφέρει νέες προοπτικές για την ενδιάμεση αξιολόγηση. Ζήτω από την Κομισιό να επιδείξει ευελιξία σε σχέση με το κανονισμό ΦΕΝΤΕΡ όταν ζητήσει ένα κράτος μέλος τα λειτουργικά ε, προγράμματα ή το εθνικό πλαίσιο αναφοράς αναθεωρηθούν θα μπορούσε η κρίση να οδηγήσει σε ορισμένες αλλαγές σχετικά με τις προτεραιότητες τι δημοσιονομικές για την κατάλληλη χρηματοδότηση των τομέων προτεραιότητας. Θα πρέπει να προωθήσουμε την ελληνική αποτελεσματικότητα στους ενεργειακούς πόρους, ε, στι υποδομές μεταφορών στην γεωργία, ε, υποδομές μεγάλου φάσματος στην Ήπεθρο, ούτως ώστε να βοηθήσουμε στην δημιουργία θέσεων εργασίας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ε, η κυρία Παλμ Χαβανόβα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σας πάνω σε περίπτωση ε, ε, ε, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, πικών της Βουλγαρίας που κατηγορούνται ότι έκαναν εγκλήματα. Ένας φοιτητής φαρμακευτικής στις 8 Ιουνίου συνελήφθη στο σπίτι του στην Σόφια και κατηγορήθηκε ότι είχε συμμετάσχει σε μια απόπειρα. Δύο μάρτυρες είπαν ότι εκείνη την εποχή ήταν στο σπίτι του και επίσης βρισκόταν και στο τοπικό σούπερ μάρκετ, πράγμα που έχει ε, το βλέπουμε στις κάμερες ε, του καταστήματος. Παρ' όλα αυτά κρατήθηκε για 70 μέρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της προφυλάκησης η αστυνομία ε, δεν θέλησε να δει τα όσα είχαν καταγράψει οι κάμερες και δεν δέχθηκε κανέναν μάρτυρα. Νομίζω ότι είναι μια περίπτωση παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων άνευ προηγουμένου που γίνεται πρακτική ρουτίνα στη Βουλγαρία. Νομίζω ότι τέτοιες προφυλακίσεις δεν δικαιολογούνται. Πρέπει να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια στο Υπουργείο Εσωτερικών της Βουλγαρίας. Κύριε Πρόεδρε, εδώ και 70 μέρες 32 ε, φυλακισμένοι Μαπούτς ε, βρίσκονται ε, σε υπεργία πίνης και κινδυνεύει η ζωή τους διότι ε, δεν έχουν δικαίωμα πρόσβαση στη γη και δεν μπορούν να υπερασπιστούν το κοινό δίκαιο. Ε, ε, οι διεθνείς συμβάσεις προβλέπουν ότι οι αυτόχθονες πρέπει να έχουν πρόσβαση στην συλλογική ιδιοκτησία στο έδαφος τους που ανήκει, ανήκει στους προγόνους τους. Στην Χιλή αυτό δεν έχει αναγνωριστεί και υπάρχουν μέτρα δυσανάλογα που έχουν ληφθεί κατά της, του πληθυσμού Μαπούτς που αντιπροσωπεύει ωστόσο 5% του πληθυσμού. Για να ε, ε, διασωθεί ο πληθυσμός Μαπούτς θα πρέπει η Χιλή να αναγνωρίσει τα δικαιώματα του πληθυσμού αυτού και τις διεκδικήσεις τους θα πρέπει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως τα Ηνωμένα Έθνη και αλλού σε διεθνείς οργανισμούς να αγωνιστούμε ώστε τα δικαιώματα των αυτοχθόνων να γίνουν σεβαστά. Τι σκοπεύετε να κάνετε κύριε Πρόεδρε για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πόρτας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από δύο χρόνια είχαμε την κατάρρευση της Lehman Brothers, η οποία ξεκίνησε ε, το κράχ της, στα χρηματιστήρια και την χρηματοπιστωτική κρίση την οποία βιώνουν ακόμα οι χώρες μας. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε έναν απολογισμό τη κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδρασε γρήγορα, ήταν σκληρή, ήταν, ε, ε, επέδειξε μεγάλη έλλειψη ευελιξία στην εφαρμογή προγράμματο, αλλά πάρα πολύ αργή σε οτιδήποτε άλλο, σε οτιδήποτε θα μπορούσε να σημαίνει κοινωνική δικαιοσύνη στην οικονομία. Μόνον αυτή την εβδομάδα το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει τα πρώτα μέτρα για την ε, χρηματοπιστωτική επιτήρηση, εποπτεία σε νέα χρόνια οι τράπεζες θα εφαρμόσουν τους κανόνες που καθορίστηκαν ε, για τα ίδια κεφάλαια. Και τα πρώτα πράγματα τα οποία έλεγαν ήταν ότι θα καταπολεμήσουμε την κερδοσκοπία, πρέπει να πάψουν να υπάρχουν η φορολογική παράδοση, θα πρέπει να υπάρχει ένα φόρο για τις ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Όλα αυτά πέρασαν στι καλένδε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν στι 29 Σεπτεμβρίου να είμαστε όλοι ενωμένοι γιατί είναι η μάχη σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπεκάλη δεν είναι εδώ. Να περάσουμε λοιπόν στην κυρία Μορβάη. Ευχαριστώ. Μπορείτε βεβαίως να καταλάβετε ότι υπάρχουν ομάδες ε, θυμάτων εγκλημάτων που υφίστανται καθημερινά σεξουαλική και σωματική βία και ηθική βία και διάφορες μορφές τρομοκρατίας, Η βία κατά των γυναικών και η βία εντός της οικογενείας ή μέσα στο ζευγάρι. Εδώ μιλάω πάντοτε για γυναίκες διότι ήρθαν σε επαφή μαζί μου και μου είπαν ότι δυστυχώς στην Ουγγαρία αυτή η σημαντική ομάδα δεν έχει επαρκή στήριξη. Όταν δηλαδή πηγαίνουν στην αστυνομία τους λέγουν ότι είναι ιδιωτικές πολλές υποθέσεις και δεν θέλουν να επέμβουν και πηγαίνουν στην ΤΑΣ ε, και τους λένε κάτε ε, ε, μην πάτε γιατί θα κρατήσουν τα παιδιά σας τότε. Οπότε θα ήθελα να κάνω μία έκκληση σε όλους τους ευρωβουλευτές να οργανωθούν και να ενισχύσουν την οργάνωση αυτή μέσω μιας συναντιάσεως για να ακουστούν τα προβλήματά τους. Ευχαριστώ. Η κυρία Κουετσέρα για ένα λεπτό. Ο κύριος Κουετσέρα. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και πάλι η ε, Πορτογαλία επλήγει από τις ε, πυρκαγιές των δασών που κατέστρεψαν πολλές ιδιοκτησίες ε, και ήταν εις βάρος του εντοπίου πληθυσμού. Είχαμε πάνω από 9.000 πυρκαγιές που είναι ο μεγαλύτερος αριθμός από το 2006. Δεδομένης της δύσκολης κατάστασης πρέπει να εξετάσουμε τις αιτίες αλλά και να επιζητήσουμε λύσεις θα χρειαστούμε προγράμματα για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτές τις πυρκαγιές και χρειαζόμαστε και υλικό και ανθρώπινο υλικό για να βοηθήσουμε τους, ε, ε, τα άτομα τα οποία έχουν πληγεί. Τον Αύγουστο είδαμε και πάλι ε, προβλήματα, ιδίως στα νησιά και υπήρχαν οι δυσκολίες που ο περιέγραψε στη Μαδέρα, χρειάζονται δηλαδή κάθε βοήθεια για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι είναι ευχάριστο ε, να ε, βλέπετε την κατάσταση εις ε, την χώρα μου διότι τα ομόλογα στην Ιρλανδία είναι σε πολύ δύσκολη θέση και γι' αυτό οι ψηφοφόροι μου ρωτούν τι γίνεται διότι υπάρχει μεγάλη κερδοσκοπία. Χαίρομαι διότι ότι προσφάτως ο ε, Επίτροπος ζήτησε να κλείσει μία Αγγλοϊρλανδική τράπεζα η οποία έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξη της χώρας μου και ε, βλέπουμε ότι υπήρχαν ε, τεράστια δάνεια και μόνο με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τη σταθερότητα θα μπορέσει να επανέλθει η ηρεμία στη χώρα μου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάτσιν έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το Σαββατοκύριακο η Σλοβενία αντιμετώπισε μεγάλες βροχές και πλημμύρες που οδήγησαν σε μεγάλες οικονομικές ζημιές. Ε, ξεχύλισαν τα ποτάμια και ε, οι πλημμύρες αυτές έσπασαν ρεκόρ 100 ετών και ε, πάρα πολλοί πνίγηκαν, πνίγηκαν μέσα στο ίδιο το αυτοκίνητό τους η Λιουγκάνα Έχουμε πάρα πολλά σπίτια, εκατοντάδες σπίτια κάτω από τα νερά. Ε, η υποδομή, η κοινοτική έχει πληγεί. Είμαστε μια μικρή χώρα, αλλά οι συνέπειες μπορούν να συγκριθούν με τις καταστροφικές συνέπειες που παρατηρήθηκαν σε μερικές χώρες της Κεντρικής Ευρώπης στην αρχή του έτους. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτές τις ανησυχίες, διότι νομίζω ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασχοληθούμε με τις συνέπειες αυτές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σόντεμπαρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην τελευταία, από την τελευταία μας ολομέλεια πάνω από 50 μητέρες από την στους Κούρδους ε, είχαν στείλει ανοιχτή επιστολή ε, στον Πρωθυπουργό των Δανών της εποχής. Είναι παράλογη η κατάσταση σε αυτήν την χώρα υποψήφια ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τιμωρούνται άτομα επειδή έστειλαν μια επιστολή σε Πρωθυπουργό χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 151 Κούρδοι ε, θα προσεχθούν στα δικαστήρια στις 2 Οκτωβρίου ε, και διάφοροι δήμαρχοι ε, όπως ο Εντεμίρ που είναι αντιπρόεδρος της οργάνωσης ΙΟΝΤΕ που υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ίσως καταδικαστεί σε ισόβια. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε, κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι παρόν για να παρακολουθήσει αυτή τη δίκη. Ευχαριστώ, κυρία Ζαμπόρσκα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είχαμε τις εκτοπίσεις και απελάσεις των Ρωμά που έδειξαν την ανικανότητα να βρεθεί μια λύση της Ένωσης ε, και βλέπουμε ότι ε, είναι το πρόβλημα επίσης ε, της εξαιρετικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Χρειάζεται αλληλεγγύη, βοήθεια, μητέρες με μικρά παιδιά απομονώθηκαν και βρεθήκαν σε τέτοια κατάσταση ώστε δεν είναι σε θέση να αλληλοβοηθηθούν. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Είναι θέμα να αρχίσουμε να συμπεριφερόμαστε σαν μια κοινότητα που φροντίζει ε, για τα άτομα, για τους ανθρώπους. Θα πρέπει να έχουμε εθελοντές για να βοηθήσουν κοινωνικά αυτά τα άτομα, τα εξαρτώμενα άτομα κοινωνικά. Ας βρούμε αυτούς τους εθελοντές για να βγούμε από αυτόν τον φαύλο κύκλο. Ευχαριστώ κύριε Μπλινκεβιτσιούτε για ένα λεπτό τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όταν το κοινοβούλιο της χώρας μου απέριψε ε, νομοθετικές τροπολογίες ε, για τη βία κατά των παιδιών, αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι οι κοινωνίες μας ε, κυριεύεται από έλλειψη ενοχής προς τους πιο ευάλωτους και στα παιδιά και δεν θέλει να προασπίσει τα δικαιώματα των παιδιών και των νέων. Για άλλη μια φορά προκύπτει η ανάγκη να διασφαλίσουμε την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Δυστυχώς οι περισσότεροι στη χώρα μου θεωρούν ότι το χαστούκι είναι πολιτιστική κληρονομιά και είναι ο καλύτερος τρόπος διαπαιδαγώγησης. Εγώ διαφωνώ κάθετα. Ε, θεωρώ ότι αυτή η πρακτική είναι αδικαιολόγητη και η βία προς ε, τα παιδιά είναι αποτρεπτική για την ε, ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών. Τα παιδιά είναι από τις πιο ευάλωτες ε, ομάδες στην κοινωνία μας και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει τα μέτρα για την καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών ε, εφαρμόζοντας δεσμευτικούς τόπους σε όλα τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να συνεργαστούν από κοινού με τα κράτη-μέλη ώστε να μην υπάρχει βία κατά των παιδιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στην πρωτοβουλία που πολλοί από εσά γνωρίζουν ήδη, αλλά που χρειάζεται περισσότερη ενίσχυση από μέρου μα. Το λεγόμενο Model European Council. Μέσω τη πρωτοβουλία αυτή, νέοι Ευρωπαίοι επιδιώκουν μια καλύτερη κατανόηση τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση χάρη στη διοργάνωση εικονική συνόδου Ολομέλεια στο Στρασβούργο σε περιόδους χαμηλής εκλογικής προσέλευσης και γενικής απάθειας είναι σημαντικό να υποστηρίζουμε και να βοηθάμε όσους ενδιαφέρονται και επιθυμούν να συμβάλλουν στη διαδικασία ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής ένωσης. γι' αυτό εν ώψη της φετινής έκδοσης του model european council σας καλώ να συναντήσετε τα μέλη των εθνικών σας αντιπροσωπιών έτσι ώστε να τους δώσουμε μια πραγματική γεύση του πώς δουλεύουμε. όσο περισσότερο προωθήσουμε αυτή την πρωτοβουλία τόσο εκείνη θα κερδίσει σε αξία για το μέλλον της Ευρώπης που οικοδομούμε εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μέλλο. Κύριε Πρόεδρε, η απόφαση του Συμβουλίου να ανοίξει την ευρωπαϊκή αγορά στην ε, κλωστοϊφαντουργία του Πακιστάν είναι λάθος. Πρόκειται για το 20% της μεταποιητικής βιομηχανίας στην Πορτογαλία. Θα χαθούν λοιπόν χιλιάδες ε, θέσεις εργασίας. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό τομέα στην Πορτογαλία, όπως είναι η αυτοκινητοβιομηχανία για τη Γερμανία, την Ιταλία ή τη Γαλλία θα ζητηθεί από αυτές τις επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν απευθείας με τις επιχειρήσεις του Πακιστάν που δεν λαμβάνουν υπόψη την κοινωνική προστασία των εργαζομένων, δεν λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντική προστασία και δεν υπάρχει καμία μέρημνα για τη χρήση συγκεκριμένων ε, επικίνδυνων πρώτων υλών. Και φυσικά η παιδική εργασία είναι ε, πραγματικότητα στο Πακιστάν. Θα ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε ότι οι επιχειρήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να ανταγωνιστούν αλλά ε, θέλουν να υπάρχει εργασία εκεί όπου παραβιάζονται όλοι οι κανόνε αγορά. Πρόκειται για μια διαμαρτυρία. Θα ήθελα να σα επιστήσω την προσοχή στο θέμα αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλι μπορέσει θα πρέπει να συζητήσει αυτό το τόσο σημαντικό θέμα για την κλωστροφαντουργία τη Ισπανία. Ευχαριστώ κύριο Σκουτάς. Η Ευρώπη σε un moment de cumpănă, în care ecoul măsurilor de austeritate se manifestă prin diferite greve. Κύριε Πρόεδρε, Βλέπουμε ότι παντού υπάρχουν ε, απεργίες στη, στα σχολεία, στις μεταφορές, στη Γαλλία, στην, ε, ε, στα σχολεία και στις μεταφορές στην Ελλάδα. Και βλέπουμε ότι όλες αυτές οι κινητοποιήσεις θα επιδεινωθούν στους επόμενους μήνες, οπότε πρέπει να έχουμε σαν στόχο την ε, οικονομική ε, ε, ανάπτυξη, την διεύρυνση της απασχολήσεως και θα πρέπει στο κέντρο της Ευρώπης να υπάρξει αλληλεγγύη. Άρα θα πρέπει να ενισχύσουμε τα κράτη-μέλη που έχουν δυσκολία για να εξέρθουν από την κρίση, για να αποφύγουμε τις πολλώσεις μεταξύ της οικονομίας των διαφόρων χωρών και για να στηρίξουμε τα κοινωνικά μέτρα αυτών των ε, πολιτικών λιτότητος. Η κυρία Φαζά. Κυρίες και κύριοι, είμαι θυμωμένη και απογοητευμένη. Αυτό πρέπει να σας πω. Και αυτό λένε οι Σλοβαίνοι όταν έγινε η πρώτη κατανομή θέσεων όχι γιατί η Σλοβίνια έχασε στην πρώτη κατανομή των θέσεων αλλά διότι 29, 29 ε, θέσεις θα καλυφθούν από τέσσερα υποψήφια κράτη και οι φιλοδοξίες των νέων κρατών είναι πιο ισχυρές από των παλιών χωρών και πάρα πολλές θέσεις καλύπτονται ακόμη από υπηκόους των παλαιών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και αυτό είναι λάθος. Πρέπει να ακούσουμε τους νέους διότι εδώ πρέπει να παίρνουμε απόφαση όλοι μαζί και θέλω να κατακρίνω το γεγονός αυτό. Δεν θέλω να υπάρξει ένα νέο σχίσμα. Πρέπει να ενωθούμε, να είμαστε ισχυροί όλοι μαζί, να έχουμε την ενωμένη φωνή των 27 χωρών και όχι μερικών εξ αυτών ο κύριος Μάτο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω για τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις τρίτες χώρες. Αναφέρθηκα στη συμφωνία με την Κολομβία και το Περού που είναι πάρα πολύ σημαντική για τις μπανάνες των Καναρίων νήσων και σήμερα θα αναφερθώ στο Μαρόκο. Εγκρίνεται σήμερα η νέα συμφωνία για την γεωργικά προϊόντα με το Μαρόκο και ε, οι ντομάτες ε, θα διευρυνθούν για όλο το χρόνο και δεν αναθεωρείται το νέο καθεστώς πληρωμών, ένα καθεστώς που ε, όπως μας είπε η Υπηρεσία Καταπολέμησης Απάτης ήταν πολύ ε, επιζήμιο για την Ισπανία, για τις περιοχές της Μούρθια, των Καναρίων Νήσων και γενικότερα για όλη την Ισπανία. Δεν είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας προστείνει μια νέα συμφωνία χωρίς εγγυήσει, χωρίς να λαμβάνονται μέτρα. Θα πρέπει να αναθεωρηθεί κατεπηγόντως το σύστημα τιμών εισαγωγή και θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το προχωρήσει χωρίς καμία καθυστέρηση. Η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως ρόλο να προσπίσει τους αγρότες. Ας το κάνει επιτέλους. Thank Ευχαριστώ. Ο κύριο Λίξφριτ δεν είναι στη θέση του. Η κυρία Πλάμ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Σήμερα θέλω να μιλήσω για τον σεβασμό του κράτους δικαίου και ε, του επαγγελματισμού στην ε, ρουμανική δημόσια διοίκηση διότι αντεκατεστάθησαν προσφάτως ορισμένοι νομάρχες και η αιτιολογία που δόθησε, δόθηκε ήταν ότι ε, είχαν αναλάβει προσωρινά τις θέσεις μέχρι ότου προκηρυχθεί διαγωνισμός. Τέλος έγινε ο διαγωνισμός και κοινοποιήθηκαν τα αποτελέσματα αρχές Οκτωβρίου 2009. Έπρεπε λοιπόν να τοποθετηθούν οι επιτυχόντες στις θέσεις, πράγμα το οποίο δεν έγινε. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι υπάρχει ε, μία κατάχρηση από το, Γερμα... από το Ρουμανικό κράτος, το οποίο θα πρέπει να σεβαστεί το κράτος δικαίου και τον επαγγελματισμό στη δημόσια διοίκηση. Ο κύριος Γιούρκ. Ευχαριστώ. ένα, ε, μία από τις ε, πρώτες ε, επιτυχίες, από τις πιο σημαντικές επιτυχίες της κοινή ευρωπαϊκής πολιτικής είναι ότι η εξωτερική υπηρεσία θα λειτουργήσει ως ο νουπο. Αλλά δεν, δεν έχει υπάρχει σωστή κατανομή των θέσεων. Από 30 θέσεις μόνο 4 πήγαν στα νέα κράτη-μέλη και δεν έγινε μία κατανομή να χώρα ε, κατά την κατάρτιση αυτού του καταλόγου θα έπρεπε να υπάρχει μία αναλογική ε, παρουσίαση και κατανομή και θα παρακαλούσαμε την κυρία Άστον στο μέλλον να σέβεται τις αναλογίες είτε πρόκειται για επικεφαλής αποστολών είτε για εντεταλμένους διότι διαφορετικά δεν μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι αυτό το σημείο είναι απλώς μία τυπική διαδικασία. Ο κύριος Μαρινέσκου δεν είναι στη θέση του και δίνω το λόγο στον κύριο Κούκαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ένα επίκαιρο θέμα. Περιμένουμε την ε, προσχώρηση της Ισλανδίας και Κροατίας που θα είναι ένα βήμα που θα, που ενθαρρύνει όσους υποστηρίζουν ε, τη διεύρυνση και συνέχισή της και αυτό θα ενθαρρύνει και άλλα ε, χώρες των Δυτικών Βαλκανίων κυρίως αυτές τις ημέρες με την οικονομική κρίση και την αυξανόμενη αβεβαιότητα στην περιοχή αυτή. Υπήρξε συμβιβασμός ανάμεσα στη Σερβία, ε, και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν ένα υιοθετήθηκε στα Ηνωμένα Έθνη σχετικά με την ανεξαρτησία του Κωσυφοπεδίου και αυτό βοηθάει την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιλύει φλέγοντα θέματα σε διάφορες περιοχές. Κυρίως σε αυτή την περιοχή η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να παίξει ένα ρόλο στο διάλογο ανάμεσα στη Σερβία και στο Κωσυφοπέδιο και αυτό θα ε, επηρεάσει σημαντικά την αξιοπιστία της. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βαλέσα. Ο κύριος Βαλέσα. Θα ήθελα να πω μερικά λόγια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 Θα μπορούσατε να ξαναρθείτε. Με συγχωρείτε, μπορείτε να ξαναρχίσετε παρακαλώ. Θέλετε να ξαναρχίσω από την αρχή. Ναι, ναι, με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος. Ναι. Θα ήθελα να πω μερικά λόγια κατά της Χούντας στη Βυρμανία ε, και της εκλογικής επιτροπής ε, η οποία δήλωσε ότι η λύση ε, είναι αυτή στην το κόμμα της Δημοκρατίας έχει ως πρόεδρο κυρία Αν Σαν που έχει λάβει το βραβείο Ζαχάροφ από αυτό το κοινοβούλιο, η οποία είναι υπέρ του διαλόγου ανάμεσα στη Χούντα και στην αντιπολίτευση και το όταν το 2000 ε, διαπραγματεύθηκε με τους ε, στρατηγούς για την απόσυρση ε, της Χούντας από την πολιτική ζωή, αλλά χωρίς καμιά επιτυχία. Οι εκλογές τον Νοέμβριο θα είναι οι πρώτες εκλογές μετά τις τελευταίες, όταν η κυρία Αγκ τοποθετήθηκε σε κατοίκον περιορισμό ε, και το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να αντιτεθεί ε, στο στρατιωτικό ε, καθεστώς στη Χούντα που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λουχάν έχει τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να δώσω προτεραιότητα ε, στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Η συνοχή κοινωνική και εδαφική είναι στόχος για την προώθηση της παιδείας, της εκπαίδευσης και των προσόντων τοπικά και περιφερειακά. Κάθε περιφέρεια μπορεί να αναβαθμιστεί εάν έχει στην επαγγελματική κατάρτιση αυτές τις διαστάσεις. Έχουμε επαγγέλματα που βρίσκονται μόνο σε ορισμένες περιοχές και που σιγά σιγά εκλείπουν διότι δεν περιλαμβάνονται στα προγράμματα εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο. Αυτό ισχύει επίσης και για τους τοπικούς ανθρώπινους πόρους διότι αν δούμε την ιστορία, την ιστορία που μεταδίδεται προφορικά, θα πρέπει τέτοια σχέδια να υποστηριχθούν χρηματικά για να υπάρξει αυτό, αυτής, ε, ο τοπικός χαρακτήρας, ο περιφερειακός χαρακτήρας που να προωθηθεί. Θα πρέπει ε, τα ταμεία, τα ευρωπαϊκά να βοηθήσουν για αυτά, εντελώ πολλά επαγγέλματα και τέχνες θα χαθούν για πάντα. Η κυρία ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ενημέρωσης για τις ε, δασοπυρκαγιές, ε, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι πορτογαλικό. Ε, χάθηκαν 150 στράματα από τις 3, μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου φέτος το καλοκαίρι. Πρόκειται για ένα τεράστιο κόστος, περίπου 75 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν περιβαλλοντικές εμπίες και κοινωνικές εμπίες και θα πρέπει να μπορέσουμε να δούμε τι πρέπει να γίνει. Ε, η αναδάσωση είναι μια πολύ αργή διαδικασία, πολύ δύσκολη και οι πυρκαγιέ κάθε χρόνο απασχολούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν δεν είναι η Πορτογαλία, είναι κάποια άλλη χώρα. Θα πρέπει λοιπόν να ε, ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τα διάφορα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουμε από το 1995 και τούδε ε, για την καταπολέμηση των πυρκαγιών. Κυρίως το ψήφισμα που είχαμε πέρσι για τις φυσικές καταστροφές ε, οι οποίες προκαλούνται από τον άνθρωπο και εγώ ήμουν και σκιώδης εισηγήτρια στην έκθεση αυτή. Ε, τα ψηφίσματα αυτά δυστυχώς ε, πολύ δύσκολα μεταφράζονται στην πράξη και δεν είναι και πολύ αποτελεσματικά τα μέτρα που λαμβάνονται. Θα πρέπει λοιπόν το ζήτημα να ξανασυζητηθεί και κάθε φορά θα, αν δεν το λύσουμε θα βρισκόμαστε εδώ να το συζητάμε. Ολοκληρώσαμε λοιπόν με τις πολλόλεπτες παρεμβάσεις.